Dear colleagues, good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της ΕΚ, τον κύριο Ντεγκίντος, πριν περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντεγκίντος. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 29ης Νοεμβρίου ε, και 1 Δεκεμβρίου στις, ε, του Φεβρουαρίου επίσης ε, και θα ήθελα να δούμε λιγάκι και να εγκρίνουμε και τις αποφάσεις των συντονιστών. Δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη συζήτηση για το Brexit οι συντονιστές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους ε, για αυτά που προσέφεραν οι Πολδοκέικο και είπαν επίσης ότι για να διευκολυνθεί η κοινοβουλευτική εργασία θα πρέπει αυτό να ζητηθεί Θα πρέπει να συμπεριληφθούν βέβαια και περισσότεροι συνομιλητές ο προϋπολογισμός του 2020 με προτεραιότητες 20 ε, Μαρτίου είναι η καταληκτική μερομηνία. ήταν ε, για να, σταθεί, να σταλεί μια συστατική επιστολή και οι συντονιστές εκλήθησαν να καταλάβουν, ε, καταβάλουν τις προτάσεις τους Επίσης η οικονομική βοήθεια, η σχετική ομάδα εργασία. Συμφωνήσαμε σε αυτήν την επιτροπή, επιτροπή με τον Επίτροπο κύριο Μοσκοβισή στο Στρασβούργο και συμφωνήσαμε και με τον κύριο Κοστέλο η Γραμματεία θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες μία συνάντηση με τον πρόεδρο της ε, ΕΚΤΕ, τον κύριο Ντράγκη, τον Ιούλιο. Όσον αφορά το θέμα του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μετά την επιστολή της 7ης Μαρτίου ε, και τον κανονισμό, αποφασίστηκε ότι οι συντονιστές θα πρέπει να τοποθετηθούν γι' αυτό το σύμφωνο ε, το χρηματοπιστωτικό. Επίσης, έγινε δεκτό ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την απόφαση των συντονιστών να μην γίνει τίποτα για το σύμφωνο σταθερότητα σε αυτή τη φάση. Γιατί το θέμα ε, θα πρέπει να ε, αποφασιστεί και να κριθεί στο πλαίσιο της Ολομέλειας. Και τέλος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, σήμερα θα ψηφίσουμε και έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία με την αναθεώρηση του πακέτου ε, της του ΙΣΕΦΕΣ στις 23 ε, Μαρτίου συμφωνήσαμε να διατηρηθεί η τρέχουσα μορφή διακυβέρνησης αλλά συμφωνήσαμε επίσης να δώσουμε την ε, δυνατότητα επιθεώρησης ε, διοικητικά στελέχη και σε εκείνους που δίνουν στοιχεία εκτός από αυτούς που είναι τοπικοί. Η Επιτροπή λοιπόν σήμερα θα ζητηθεί άποψή τη για την συμφωνία σχετικά με το Φισκάλις αυτό συμφωνήθηκε στις 21 Μαρτίου. Οι συνομοθέτες συμφώνησαν να συνεχιστεί το επιτυχημένο πρόγραμμα φυσκάλης και κατά την επόμενη περίοδο για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ε, να υπάρξει επιλογή των εξωτερικών συμβούλων και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, ε, συμφωνήθηκε επίση ότι θα πρέπει να προσκληθούν εμπειρογνώμονε από τρίτε χώρε, κυρίω από λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, και να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε στο πρόγραμμα να, να προβλεφθούν νέες εξελίξεις. Δεν συμφωνήθηκε, δεν επιτεύχθηκε η συμφωνία στον προπολογισμό με βάση τη κατεξοδότηση και τι ε, ε, εξοδοτημένε πράξει. Η Επιτροπή θα κληθεί να τοποθετεί και πάλι σε αυτή την μερική προσωρινή συμφωνία. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Ντεγκίντος, αλλά είχα να κάνω όλες αυτές τις ανακοινώσεις που ήταν αρκετά μακροσκελής. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 5 της μερίσιας διάταξης. Καλωσορίζουμε και πάλι τον κύριο Ντεγκίντος, ο οποίος είναι παρόν για να μας παρουσιάσει την η έκθεση της ΕΚΤΕ για το 2018. Και η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε σε 22 επίσημες ε, γλώσσες σήμερα στις 3 η ώρα καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες, το περιβάλλον του 2018 συμπεριλαμβανομένης νομισματικής πολιτικής, ε, την αγορά για τις ε, πληρωμές και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ε, τα νομίσματα, στατιστικές έρευνες, νομικές δραστηριότητες, εξωτερική συνεργασία. Η ΕΚΤ επίσης δημοσίευσε την αντίδρασή της στις προτάσεις και τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά της για την ΕΚΤ το 2017. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ χρήσιμη και σημαντική συζήτηση και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο για τις εισαγωγικέ παρατηρήσεις στον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, κυρίες και κύριοι, ε, με μεγάλη τιμή, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ήρθα εδώ για πρώτη φορά στην Επιτροπή σας ως ε, Αντιπρόεδρος της ε, ΕΚΤ και χαίρομαι που θα παρουσιάσω την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2018. Η ετήσια έκθεση είναι το βασικό προϊόν λογοδοσίας της ΕΚΤ, όπως προβλέπεται από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια πολύ πέρα από τις απαιτήσει ε, των συνθήκων. Τμήμα αυτής της υγιούς και επικοδομητικής ε, σχέσης και με βάση τα ιωθώτα δημοσιεύουμε σήμερα ε, μία γραπτή έκθεση για το ψήφισμα ε, το δικό σας για την προηγούμενη ετήσια έκθεση. Μεταξύ άλλων, ε, μιλάμε για τα συνολικά ποσά των κερδών που έγιναν χάρη στο πρόγραμμα κινητών αξιών, όπως ζήτησε και το ψήφισμά σας, που ζήτησε, λένε, να δημοσιευθούν. Θα συζητήσω τι αποφάσει νομισματική πολιτική ε, για το 2018 και την επίπτωσή του στην οικονομία τη Ευρωζώνη. Ε, Όπω συμφωνήθηκε στην ετήσια έκθεση, ε, χρειάζονται επαρκή νομισματικά κίνητρα, ούτω ώστε να συγκλίνει ο πληθωρισμό στα επίπεδα του 2% κοντά, αλλά κάτω από το 2% μεσοπρόθεσμα. Επίση, θα σα δώσω μία επισκόπηση των αποφάσεων που έλαβε το Δουσού τη ΕΚΤ τη 7 Μαρτίου καθώ και βασικά στοιχεία τη οικονομική ατζέντα ε, στα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς προχωρούμε στο τέλος της ε, κοινοβουλευτικής θητείας και αυτού του ε, νομοθετικού κύκλου. Η, τα μέτρα νομισματική πολιτική συνεισφέρουν σε πολύ καλέ ε, οικονομικέ συνθήκε, υποστηρίζοντα την επέκταση τη ευρωζώνη σε όλο το 18. Ε, τα ποσοστά δανεισμού για τα νοικοκυριά και τι εταιρείε τη Ευρωζώνης ε, παραμένουν κοντά στα ιστορικά ελάχιστα επίπεδα και η ανάπτυξη του όγκου δανεισμού των τραπεζών συνεχίζουν την ανωδική του στάση που παρατηρήθηκε από τι αρχέ του 2014. Οι εταιρείε ειδικά υποφελήθηκαν από την αγορά ομολόγων ε, στο μη τραπεζικό τομέα, του ε, CSPP. Το CSPP ε, εξασφαλίζει χρηματοδότηση ε, που στα πλαίσια της αγοράς σε πιο χαμηλές ε, και προσιτές Ε, απελευθερώνει ε, δυνατότητα δανεισμού για, στους ισολογισμούς τραπεζών και έχει ε, θετική επίπτωση στην προσφορά πίστοσης, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νομισματική πολιτική υποστήριξε την εσωτερική ζήτηση και η ανάπτυξη ήταν με μέτρια το 2018. Το ΑΕΠ έφτασε, αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το 2,4% το 2017. Αυτό οφείλεται σε ε, πιο αδύναμες τάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και σε κάποιους προσω... Ε, συγκυριακούς ε, παράγοντες τόσο σε εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα βασικό στοιχείο είναι η μετάβαση στις, στα νέα πρότυπα εκπομπών για τα αυτοκίνητα που προκάλεσε κάποια συμφόρηση στην παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ε, τα μέτρα για τον λανθάνοντα ε, πληθωρισμό παρέμειναν γενικά με σε όλο το 18, αλλά ο κίνδυνο από πληθωρισμού ε, σχεδόν εξαφανίστηκε και ο πληθωρισμός είναι σε ανωδική τάση. Η δύναμη της εσωτερικής οικονομίας στηρίχθηκε από την κατάλληλη νομισματική πολιτική και τις πιο σφιχτές αγορές εργατικού δυναμικού που σπρώχνουν προς τα πάνω τους ε, μισθούς ε, και υποστηρίζουν την υποστήριξη, ε, την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμό είναι σε φάση σύγκληση σε επίπεδα κάτω αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Έχουμε αποφασίσει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αγορά περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του 2018. Ενισχύουμε την καθοδήγησή μας σε ό,τι αφορά διάφορα στοιχεία τα επιτόκια ε, είναι αυτά που θέλουμε. Ε, ο συνδυασμός των δύο στοιχείων ε, μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα υπάρξει σταθερότητα των τιμών. Επίσης, ε, η πολιτική μας για τα επιτόκια έχει ενισχυθεί από επανεπενδύσεις ε, ουσιαστικού ποσοστού ε, όλων των αγοραστέντων περιουσιακών στοιχείων. Η επανεπένδυση θα διατηρηθεί, θα διατηρήσει το μέγεθος των χαρτοφυλακίων κινητών αξιών και μαζί με την ε, καθοδήγηση που δίνουμε για την, ε, τις επανεπενδύσεις θα υποστηρίξουμε τις ε, θετικές οικονομικές συνθήκες. Από τα μισά του 2018 ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης Ευρωζώνης ήταν μέτριο παθής, αλλά καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι απογοητευτικός στις αρχές του 2019 και αυτό σημαίνει ότι η μέτρη αυτή ανάπτυξη θα συνεχιστεί το 2019. Ε, η επίπτωση των ε, εσωτερικών παραγόντων ε, μειώνουν τις τάσεις ανάπτυξης και η παγκόσμια οικονομία δεν υποστηρίζει γενικά και τη δική μας οικονομία. Υπάρχουν αβεβαιότητες, ειδικά σε γεωπολιτικό επίπεδο, ε, υπάρχουν απειλές προστατευτισμού, ε, υπάρχουν προβλήματα στις αναδυόμενες αγορές και άρα ε, αυτό υποσκάπτει τις οικονομικές τάσεις ανάπτυξης. Η τελευταία προβλέψη του προσωπικού μας για την Ευρωζώνη έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω το 19 και θεωρούμε θα φτάσει στο 1,1. Επίσης, η επίπτωση αρνητικών παραγόντων επηρεάζει την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αναμένεται στο, να φτάσει στο 1,5% το 2021 ε, και δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Οι θετικές ε, οικονομικές προϋποθέσεις, ε, κέρδη στην απασχόληση, αύξηση των μισθών κτλ. Ε, θα οδηγήσουν σε αύξηση συνολικά της παγκόσμιας δραστηριότητα και θα υποστηρίξουν την ε, επέκταση της Ευρωζώνης. Όμως η ασθενέστερη ανάπτυξη ε, θα αφήσει το σημάδι τη στι ε, πιέσει των εσωτερικές πιέσεις τιμών και θα μειώσει την ε, προσαρμογή του πληθωρισμού σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ο λανθάνο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι αρκετά μετριοπαθής και οι προβλέψεις του προσωπικού μας θεωρούν ότι θα μειωθεί η τάση του συνολικού πληθωρισμού, η οποία τώρα προβλέπεται να φτάσει στο 1,6 στο τέλος του 2021. Επομένως, ε, θα πρέπει να κάνουμε ουσιαστικέ ε, προσαρμογές στο μισματικής πολιτικής. Στη συνάντηση του Μαρτίου αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε ε, τις, ε, τους προσανατολισμούς μας, τις, τις προβλέψεις μας. Η, επίσης, ε, είναι θετικές οι τάσεις ε, δανεισμού των τραπεζών, ε, αλλά οι αδύναμες προοπτικές μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες χορήγηση πίστοση σε επιχειρήσει και νοικοκυριά. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τι συνθήκε δανεισμού των τραπεζών, εξασφαλίζοντα την επαναχρηματοδότηση των τραπεζών λόγω της, των τραπεζικών ομολόγων που φτάσουν που φτάνουν σε ορίμανση και των εναπομείναντων TLTRO ε, που δεν θα πρέπει να υποσκάψουν μισματική πολιτική. Γι' αυτό ξεκινήσαμε το TLTRO 3 με μια σειρά από τριμηνιαίους ε, μακροπρόθεσμους στόχους επαναχρηματοδότησης ξεκίνησε το, που, ξεκίνησε το 19, που θα ξεκινήσει μάλλον το 19 και θα τελειώσει το 21 ε, με διάρκεια δύο ετών κάθε φορά. Οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να δανειστούν ε, στο 30% ε, του των αποθεμάτων των επιλέξιμων δανείων σε ποσοστό α, σε ένα επιτόκιο τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένο καθ' όλη τη διάρκεια της ε, επιχείρησης αυτής. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι όλο και πιο προβληματική και αυτό απεικονίζεται ε, στους δείκτες ε, συστημικού στρες. Η ανάλυση της ECB τονίζει ότι κάποιες εξελίξεις υποστηρίζουν την οικονομική σταθερότητα και υπάρχει μια οικονομική ανάπτυξη όλο και η οποία συνεχίζεται και βελτιώνεται η ανθεκτικότητα των τραπεζών. Όμως, ε, γενικά οι δραστηριότητες ε, ε, που ενέχουν κίνδυνο σε κάποιες χρηματαγορές αντικατοπτρίζουν γενικά, οδηγούν μάλλον σε χαμηλά premium κινδύνου. Η απουσία σαφήνειας ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του Brexit συνεισφέρει σε υψηλότερη πολιτική αστάθεια. Χάρη στις προετοιμασίες που έγιναν από τις δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, ε, το σενάριο του no deal ε, δημιουργεί βέβαια κινδύνου, αλλά που μπορούμε να του διαχειριστούμε στην Ευρωζώνη και να μην υπάρξει πρόβλημα στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια σημεία ευαισθησία ε, και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αρνητικέ επιπτώσει αν του συνδυάσουμε με κινδύνου που επηρεάζουν τι προοπτικέ τη Ευρωζώνη. αυτή την. Nevertheless, European banks can... Ε, πολλές από τις μεταρρυθμίσεις ε, ωστόσο οι οποίες ε, οδήγησαν στην διεθνή κρίση έχουν τώρα ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες ακόμα δεν αξιοποιούν πλήρως τα ωφέλη που μπορεί να τους αποφέρει η ενιαία τραπεζική αγορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες έτσι ώστε να έχουμε πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές ταυτόχρονα ενισχύοντας το κανονιστικό μας πλαίσιο και για το μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Και γι' αυτόν τον λόγο η ολοκλήρωση της τραπεζικής Ευρωπαϊκή Ένωση και ενίσχυση των κεφαλαίων αγορών θα ε, συνεχίσουν να έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά το πλαίσιο τη νέα βουλευτική ε, θητεία. Όπω ε, αναφέρουμε και στην ετήσια έκθεση, η ΕΚΟΤΟΥ το 2018 συνέχισε να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικέ συμβουλέ σε αυτό το τομέα και στου επόμενου μήνε, στο πλαίσιο δηλαδή τη προεκλογική αν περίοδου, υπάρχει μια τέλεια δυνατότητα ούτω ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ολοκληρώσουμε τι μεταρρυθμίσει που ξεκινήσει. Μια γνήσια ε, ένωση χρηματοπιστωτική, δηλαδή των αγορών και μια πλήρη τραπεζική ένωση θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να ε, λειτουργήσει καλύτερα οικονομική και νομισματική έννοια. Ε, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πιο ολοκληρωμένε αγορέ ε, και ένα καλύτερο τρόπο τη κοινή διαχείριση κινδύνου που αποτελεί βέβαια και το μειονέκτημα τη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τι ΗΠΑ. Και στο θεσμικό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το, ε, και το κοινό ταμείο έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη αντοχή του, της τραπεζικής μας ένωσης. Το σύστημα του ευρώ θα πρέπει επίσης να παίξει το ρόλο του ως καταλήτης για την, ε, να επιφέρει αλλαγή και την ενίσχυση της ε, εναρμόνισης των προτύπων της αγοράς. Προκειμένου να διευκολύνουμε την, ε, την πανευρωπαϊκή εμβέλεια των ε, άμεσων πληρωμών το 2018 το Νοέμβριο το Ευρωσύστημα, το Eurosystem ξεκίνησε μια καινοτόμα υπηρεσία το Target Instant Payment Settlement. Αυτά λοιπόν τα tips επιτρέπουν στους ε, ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις να προβαίνουν στην, σε τραπεζικές μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικές πληρωμές σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ε, ε, αυτέ οι καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και η ολοκλήρωση τη αγορά θα πρέπει να υποστηριχθούν και από τι κατάλληλε πολιτικέ σε άλλου τομεί. Ε, για, παράδειγμα, ε, πλήρη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και πιο αποτελεσματικό συντονισμό των οικονομικών πολιτιμών, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αντοχή τη ζώνη του ευρώ και να δημιουργήσουμε αξιοπιστία, εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ολοκλήρωση. Και ταυτόχρονα, βέβαια, τα θεσμικά θεμέλια τη Οικονομική και Ένωση θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε από τη μία πλευρά ε, την διαχείριση και την ε, επιχειρησιακή ικανότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, σεβόμενη πλήρω την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα θωρακίσουμε καλύτερα τα μέλη τη Ευρωζώνη από κλειδονισμού. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία ενό δημοσιονομικού εργαλείου για την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα τη ζώνη του ευρώ θα συμβάλλει στην ενίσχυση τη ζώνη του ευρώ, στην περισσότερη αντοχή τη και των κρατών μελών τη. Ε, να ολοκληρώσω όμω. Καθώ λοιπόν ολοκληρώνουμε, φτάνουμε στο τέλο αυτή τη βουλευτική θετία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, ε, αυτά τα δύο δηλαδή θεσμικά όργανα Επιτροπή με την ε, Τράπεζα, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν ήταν εύκολη η περίοδο στην οποία διανύσαμε και οι πολίτε μα δικαίω αξίωσαν να υπάρξουν αποτελεσματικέ και απτέ λύσει στι οικονομικέ και χρηματοπιστωτικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Εσεί Εσείς έχετε παίξει έναν ζωτικό ρόλο έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι προσδοκίε των πολιτών μα και για να διασφαλίσετε ακριβώ το ότι είναι υπόλογο για τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα και ταυτόχρονα εσεί ω συνομοθέτε ε, σχεδιάσατε και εγκρίνετε τι μεταρρυθμίσει οι οποίε έχουν επιτρέψει στην Ένωση να είναι ισχυρότερη σήμερα. Γνωρίζετε βέβαια ότι η μεταρρύθμιση, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι είναι μια συνεχή προσπάθεια για τα ωφέλη από αυτέ τι ε, με προσπάθειε που έχουμε κάνει ε, δεν είναι πάντοτε πολύ ορατά. Ωστόσο, όπω φαίνεται και από το Ευρωβαρόμετρο, ε, η ε, υποστήριξη του κενού προ το ευρώ το 2018 έφτασε το 75%. Άρα λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την άγουσα που, έχουμε, που ακολουθούμε ήδη έτσι ώστε να έχουμε μια πιο βαθιά και πιο ευρία οικονομική και νομισματική ένωση. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντεγκίντο. Πρώτα απ' όλα βεβαίω θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που κάνει η ΕΚΤ και προφανώς ε, λαμβάνονται υπόψη οικονομική προοπτική τα τελευταία στοιχεία και θεωρώ ότι η τελευταία απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ιδιαίτερα σοφή και γι' αυτό το λόγο προσβλέπουμε και στην επόμενη απόφαση τον επόμενο μήνα για να αντιμετωπιστεί αυτή η υφεσιακή τάση την οποία διαπιστώνουμε στις ε, ευρωπαϊκές οικονομίες. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπατε για την ε, μεταρρύθμιση της ε, νομισματικής ζώνης. Προφανώς και υποστηρίζω πλήρως και αναβιφύλακτα όλα αυτά τα οποία είπατε και κυρίως όσον αφορά τα δημοσιονομικά εργαλεία. Μερικοί από εμάς ε, είναι περισσότερο φιλόδοξοι από την είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τόσο εδώ όσο και στην ε, ΕΚΤ και στα κράτη-μέλη. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους ε, θεσμούς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε Εσείς είπατε ότι ήρθατε εδώ πρώτη φορά, εγώ το είχα μπερδέψει και είχα μπερδευτεί με την ακρόαση. Πράγματι, με αυτή την ιδιότητα και σε αυτό το πλαίσιο είσαστε εδώ πρώτη φορά. Ευχαριστούμε την ΕΚΤ για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Νομίζω είχαμε πολύ καλή συνεργασία για να βελτιώσουμε το διάλογο και για να στηρίξουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προφανώς και είναι καθοριστική σημασία. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα βελτιώσει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα καλή σχέση. Ας περάσουμε τώρα στα μέλη μας και ο πρώτος που έχει δει το λόγο είναι ο κύριος Λάγκεν. Παρακαλώ κύριε Λάγκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεγκίντος. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην πρώτη σας ε, παρουσία και παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι το βρίσκω λιγάκι απογοητευτικό το ότι εδώ στην αίθουσα είναι παρόνες μόνο 7 βουλευτές τη στιγμή που εσείς παρουσιάζετε την πρώτη σας ετήσια έκθεση. Αυτό όμως ίσως να οφείλεται στο ότι σήμερα είναι Δευτέρα, τελειώνει και η θητεία. Παρόλα αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ετήσια έκθεση με τον πρόεδρο της ΕΚΤ και με διάφορους ε, διευθυντές. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει πάρα πολλά θέματα. Εγώ θέλω να θίξω τρία. Το ένα είναι το ποσοστό του πληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία σήμερα αναφέρει ότι σε όλη την Ευρώπη κατά 1,4 μειώθηκε ο πληθωρισμός και παράλληλα ο ρυθμός της ανεργίας είναι ο χαμηλότερος από το 2008. Άρα δηλαδή αυτά είναι ιδιαίτερα ε, θετικές εξελίξεις. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό του πληθωρισμού, το ποσοστό αυτό τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό ήταν ε, συνάρτηση της ενεργειακής κρίσης ε, και της ε, ψηφιοποίησης, η οποία και με, την ίδια, την, με τον ίδιο τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τάπεζας είναι κάτω του 2%. Τι θα γίνει όμως αν πέσει περισσότερο αυτό το ποσοστό. Με αυτές τις εξελίξεις των τιμών δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει νομισματική πολιτική, πολιτική και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τον βασικό πληθωρισμό εάν αφαιρέσει κανείς τις εποχικές τιμέ και τις ενεργειακές τιμέ. Το δεύτερο που θέλω να πω, η ΕΚΤ είπε ότι νέα μέτρα ή ένα πρόγραμμα αγορά ομολόγων, ότι αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Γίνεται λόγο αυτή τη στιγμή για τα αρνητικά επιτόκια των τραπεζών. Και ρωτώ, σε ποια δεσμή μέτρων θα μπορούσαν τα αρνητικά επιτόκια να προκαλέσουν σημαντικές αναδιορθώσεις στις τράπεζες αν πραγματικά όλα αυτά που έχουν λεχθεί λάβουν, ε, εφαρμοστούν στην πράξη. Το τρίτο, η Τραπεζική Ένωση, η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Γνωρίζουμε ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρχαν ιδιαίτερα έντονες επιφυλάξεις ε, όσον αφορά τις αρχικές επιφυλάξεις για την ε, ε, εξασφάλιση των καταθέσεων. Και ισχύουν να υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι κάνετε στο, στην επόμενη θητεία με την ε, εξασφάλιση των καταθέσεων. Ε, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, ορισμένα τα οποία είναι κατηγορηματικά αντίθετα σε αυτές τις εγγύησεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκε. Νομίζω ότι τρία πράγματα ρωτήσατε. Πρώτον για τον πληθωρισμό. Δεύτερον για τα αρνητικά επιτόκια και για τις επιπτώσεις των ερνητικών επιτοκίων στις τράπεζες και τρίτον τι θα γίνει με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης του συστήματος ΙΝΤΙΣ. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ ε, σε αυτά τα οποία μας είπατε και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον πληθωρισμό. Σήμερα λοιπόν με βάση τα τελευταία στοιχεία και δημοσιεύτηκαν σήμερα πρόκειται για τα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό του Μαρτίου. Ε, θα είδατε ότι το ποσοστό του πληθωρισμού ανέρχεται σε 1,4%. Ο βασικός πληθωρισμός είναι 1,8%. Όσον αφορά την μείωση αυτή του 1,4% αυτό προέκυψε λόγω της εξέλιξης ε, των ενεργειακών τιμών, όπως είπατε βέβαια και εσείς. Είδαμε όμως και μια επιτάχυνση του βασικού πληθωρισμού, ο οποίος ήταν περίπου στο 1%, δηλαδή κάτι πάνω από το 1% ε, σε σχέση με τους 3 ε, με 5 μήνες. Τώρα όμως βλέπουμε μια πτώση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με τον βασικό πληθωρισμό. Νομίζω το βασικότερο θέμα σε σχέση με αυτόν τον πληθωρισμό είναι ότι έχουμε ύφεση της οικονομίας. Αυτή η ύφεσιακή τάση αρχίζει να έχει επιπτώσεις στο βασικό πληθωρισμό. Παράλληλα όμως υπάρχουν και δύο άλλοι παράγοντες που κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να έχουν θετικές επιπτώσεις στο βασικό πληθωρισμό κατά τα επόμενα τρίμηνα. Το ένα είναι η στρατηγική μας, η νομισματική και το δεύτερο, το είπατε κι εσείς, ε, το θέμα της απασχόλησης. Η ανεργία είναι πολύ χαμηλή, 9 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας προέκυψαν από το τέλος της κρίσης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και αύξηση των μισθών. Οι μισθοί αυξάνονται κατά 2,5% σε ορισμένε ε, χώρε ακόμα περισσότερο, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία. Εκεί οι συνθήκε εργασία είναι διαφορετικέ από τι άλλε χώρε ευρωζώνης. Όμω υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Αυτή η εξέλιξη των μισθών γιατί δεν έχει άμεση επιπτώσεις στις τιμές λιανικής. Γιατί δεν μετακυλείται αυτή η εξέλιξη από τους μισθούς στον πληθωρισμό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να εξηγήσουμε. Ίσως ε, να έχει αλλάξει η διάρθρωση των αγορών. Ίσως ε, να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στο διαδίκτυο, στην ψηφιακή οικονομία. Ίσως αυτά να επηρεάζουν τον πληθωρισμό περισσότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να εξτάσουμε πολύ προσεκτικά. Είπα και στις αρχικές μου παρατηρήσεις ότι εμείς θέλουμε να προσαρμόσουμε τη νομισματική μας πολιτική, να είμαστε ανοιχτοί, έχουμε λάβει μέτρα και όπως γνωρίζετε υπάρχει το περίφημο toolkit ε, της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής, αυτό το εργαλείο και είμαστε πεπισμένοι ότι με αυτά που προβλέπουμε για το δεύτερο εξάμεινο σε σχέση με τον πληθωρισμό και σε σχέση με τις ενεργειακές τιμές, αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά βάσει όλων αυτών των προβλέψεων θα υπάρξει ανάκαμψη και αυτό θα μας βοηθήσει έτσι ώστε ο βασικός πληθωρισμός να πλησιάσει το στόχο μας που είναι λίγο κάτω από το 2%. Το δεύτερο ερώτημα που θέσετε και είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα των αρνητικών επιτοκίων. Οι επιπτώσεις που έχουν τα αρνητικά επιτόκια στις τράπεζες. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι τα αρνητικά επιτόκια είναι πολύ σημαντικά για να προάγει κανείς την οικονομική δραστηριότητα. Και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία τρία έτη πριν από την υφεσιακή τάση που αρχίσαμε να διαπιστώνουμε στις αρχές του 2018, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κερδοφορία των τραπεζών. Τώρα λοιπόν διαπιστώνεται μία ύφεση, αλλά η χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι ξεπερνάει τις επιπτώσεις που θα μπορούσε κανείς να αποδώσει στα αρνητικά επιτόκια. Η χαμηλή κερδοφορία των ε, τραπεζών στην Ευρώπη είναι διαρθρωτική. Παραδείγματος χάρη, τα επιχειρηματικά δάνεια. Έχουμε σημειώσει εκεί κάποια πρόοδο, αλλά δεν είναι ικανοποιητική. Δεν φτάνουν αυτά τα δάνεια. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της αποτελεσματικότητας ε, σε σχέση με το κόστος. Ε, ο λόγος αυτός ε, στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, νομίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές τράπεζες. Δηλαδή, ο τραπεζικός τομέας εκεί υπάρχει κάποια υπερβολή στον τραπεζικό τομέα και ως εκ τούτου οι τράπεζες θα έπρεπε να προσπαθήσουν να περιορίσουν αυτό το πλεόνασμα. Αυτοί είναι δύο βασικοί παράγοντες. Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με την εξυγίανση, με τον περιορισμό, όπως σας είπα, του πλεονάσματος, του τραπεζικού πλεονάσματος υπάρχουν κάποιες σχετικές έρευνες που διεξάγουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων που βιώσαμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό θα συνεχιστεί να υπάρχει στην Ευρωζώνη. Τέλος, όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, για μας αυτό το θέμα είναι καθοριστική σημασίας. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα IDC ε, είναι ένα ορόσημο, είναι ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης, το χρειαζόμαστε απολύτως. Βεβαίως και η συζήτηση δεν είναι εύκολη, γιατί πρέπει να εξετάζουμε την μείωση κινδύνων και την αμοιβεποίηση, όπως αποκαλείται, των κινδύνων. Αυτά τα δύο παράλληλα Πάντως ε, το θέμα με το πρόγραμμα IDs είναι ότι θα είναι δύσκολο αν ε, δεν ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Άλλο στοιχείο είναι η ολοκλήρωση της, ε, των κεφαλαίων αγορών Οι αποφάσεις ε, για την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαγορών, οι αποφάσεις ε, θα πρέπει να ληφθούν βεβαίως ε, εφόσον θα υπάρχουν τα απαραίτητα δημοσιονομικά εργαλεία για να λειτουργήσουν αντικυκλικά. Ευχαριστώ. Η Περόν Μπερές από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για την δημοσιονομική δυνατότητα που έχουμε, το αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Μιλάμε... Ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε μιλήσει με πολύ έντονο ύφο ε, και είχε πει ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει να προχωρήσουμε και ότι χρειαζόμαστε ε, ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε, διαφορετικό, να υπάρχει μια καλή ισορροπία στη διακυβέρνηση. Προφανώς τα πράγματα δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε στο Συμβούλιο. Βλέπουμε ότι ακόμα και για την πρόταση της Κομισιόν, η οποία θεωρήθηκε δειλή, αλλά που τουλάχιστον είχε την εξής, το εξή πλεονέκτημα. Ασχολούνταν με την ε, σημασία της σταθεροποίησης της Ευρωζώνης. Κινδυνεύει να χαθεί στους ε, δεδάλους των συζητήσεων των, ε, του Συμβουλίου εσείς περιγράψατε το τραπέζι, το, συγγνώμη, το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η νομισματική πολιτική ως εξή. Ότι υπάρχουν κίνδυνοι ε, που συνδέονται με το εμπόριο, ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την όλο ένα και μεγαλύτερη πιθανότητα ενός Brexit και το πολιτικό μήνυμα που περνάει μέσα από αυτή την ε, ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, τι μήνυμα στέλνετε στον, ε, στους Ευρωπαίους νομοθέτες, ποιο είναι το πλαίσιο που χρειάζεστε ούτω ώστε η νομισματική πολιτική να παίξει σταθεροποιητικό και αποτελεσματικό ρόλο. Διότι αυτό επιδιώκουμε με αυτήν. Το πρώτο μήνυμα που θέλω να διαμηνήσω προσωπικά αφορά το εξής, ότι νομισματική πολιτική δεν είναι και τόσο παντοδύναμη. Είναι τμήμα της οικονομικής πολιτικής, ενός μείγματος οικονομικής πολιτικής. Αλλά η δημοσιονομική πολιτική παίζει ένα σημαντικό ρόλο και αυτή σίγουρα. Στο παρελθόν Μερικές φορές είχαμε την αντίληψη ότι η νομισματική πολιτική ήταν το μόνο διαθέσιμο εργαλείο για να μας ε, βγάλει από την κρίση. Η ΕΚΤ το χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο και έχουμε δει καλά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι το μόνο εργαλείο διαθέσιμο. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία της οικονομικής πολιτικής που είναι σημαντικά. Αναφέρατε ρητά την δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η δημοσιονομική πολιτική σε εθνικό επίπεδο, τι κάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις, ότι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αυτό είναι σημαντικό. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι η δημοσιονομική θέση κάθε χώρας ε, δεν είναι ίδια, είναι διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν κάποιε χώρε που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το περιθώριο, ούτω ώστε να ενισχύσουν την ε, οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν άλλε χώρε που έχουν υψηλή χρέωση, υψηλό χρέο. Ε, πολύ υψηλό λόγο δημοσίου χρέου και επομένω το δημοσιονομικό αυτό περιθώριο είναι πολύ πιο περιορισμένο. Αλλά νομίζω αν θέλετε τέλο πάντων την προσωπική μου γνώμη, για να έχουμε μια ενοποιημένη άποψη για την ε, κατάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, στηρίζουμε πλήρως αυτή την πρόταση του να έχουμε ένα δημοσιονομικό ενοποιημένο εργαλείο για την Ευρωζώνη, το οποίο θα έχει όχι μόνο στόχους ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά θα πρέπει να είναι εργαλείο σταθεροποίησης σε περίπτωση που έχουμε ασύμετρα σοκ, τα οποία επηρεάσουν τμήμα της Ευρωζώνης ή ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός περιθωρίου που έχουν ορισμένα κράτη-μέλη και τη δυνατότητα κατά συνέπεια ε, να έχουν περισσότερο επεκτατική νομισματική πολιτική μαζί με την ύπαρξη της αντικυκλικής δημοσιονομικής ε, δυνατότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης πιστεύω ακράδαντα τι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Πιστεύω ότι χρειάζονται ούτω ώστε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας μεσοπρόθεσμα και παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανές η νομισματική πολιτική δεν είναι το μόνο εργαλείο, θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε με δημοσιονομική πολιτική και διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε το σωστό μείγμα πολιτικής για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Ε, Ραμόν... Ευχαριστούμε. Ραμόν Τρεμόζε τώρα. Grazie, Presidente. Signor De Guindos. Καλησπέρα, κύριε Δεγκίντο. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Καταρχάς, το θέμα της διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως ξέρετε, στο Κοινοβούλιο και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, οι Ευρωβουλευτέ πιέζαμε για να δημοσιεύονται τα πρακτικά του προγράμματος Target 2. Και Πιέσαμε επίσης ε, τα πρακτικά των, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δημόσια. Τώρα, 40 βουλευτές δημοσία ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα να δημοσιοποιηθούν τα νούμερα των επιχειρήσεων και τα ονόματα των επιχειρήσεων που εποφελούνται από την αγορά χρέους ε, από πλευράς ορισμένων κεντρικών τραπεζών. Βεβαίω τώρα υπάρχουν και νέα προγράμματα προ αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να ξέρουμε τα ονόματα, τι ποσότητε, ε, τι ημερομηνίε, όλα. Δεύτερον, στον ευρωπαϊκό τύπο μιλάμε για πιθανέ συγχωνεύσει τραπεζών. Στη Γερμανία, η Deutsche Bank με το Commerce Bank. Επίση, το ΜΑΚΕ μπορεί να συγχωνευτεί με μια άλλη τράπεζα. Και τώρα υπάρχει, ε, υπάρχει μια ερώτηση για πλεονάζον δυναμικό στην ΕΚΤ. Θα ήθελα στοιχεία συγκεκριμένα για αυτά τα θέματα. Και τέλος, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που για μένα με απασχολεί με μανία. Το συζητάμε από καιρούς καιρών στην Επιτροπή μας. Στις 21 Νοεμβρίου του 2017 έθεσα τέτοια ερώτηση και εσείς απαντήσατε και αποδίδατε την αιτία αυτών των δανείων στη μη πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές. Late Payments Directive. Ε, στην Ισπανία, ας πούμε, δεν υπάρχει ένας κανονισμός ε, κυρώσει, με κυρώσεις για τις πολυεθνικές, ας πούμε, ε, οι οποίες μπορεί να πέρασουν και δύο χρόνια για να πληρώσουν, ας πούμε, ε, τα τιμολόγια στις α, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, προς τις, τις οποίες χρησιμοποιούν ως υπεργολάβους. Επίσης, επί πολλά χρόνια υπάρχουν εταιρείε οι οποίες δεν πλήρωναν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούσαν ως υπεργολάβους. Επί χρόνια, στη Δανία ας πούμε, ε, υπήρχε ε, μαζική ανεργία το 2010 γιατί αυτές οι εταιρείε φαλήρισαν. έτσι, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί, να εισκύψει ε, μία ευνίδια κρίση ε, και να μπορεί να, να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρεμόσα. Θέσατε τρία πολύ ευστοχά ζητήματα. Καταρχήν ε, τη διαφάνεια. Το δεύτερο ήταν ε, το ζήτημα της δυνατότητας συγχωνεύσεων γενικότερα στον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης παρόντια και βέβαια το τρίτο ζήτημα που θέσατε είναι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την καθυστερημένη αποπληρωμή τους. Θα ξεκινήσω με αυτό το τελευταίο ζήτημα. Αυτές λοιπόν οι καθυστερημένες αποπληρωμένε. Είναι κάτι το οποίο ε, βέβαια είναι ατυχε. Αλλά ε, ορισμένες φορές όπως είπατε συχνά το πρόβλημα ε, ε, δεν έγκυται στο ότι ακριβώς ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επιβάλλουν άδικους αν θέλετε τροβαρείς όρους στις μικρότερες επιχειρήσεις. Είναι το ότι γενικά γίνεται πληρωμία αλλά καθυστερημένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει εθνική νομοθεσία η οποία ακριβώς θα αποτρέπει την εμφάνιση τέτοιου είδους καταστάσεων. Γιατί όπως είπατε κι εσείς Ε, σε περίπτωση επιβράνθησης της οικονομίας, όταν υπάρξει ένα τέτοιο πιστοτικό crunch, όπως λέγεται ένα credit crunch, όπως εκείνο που σημειώθηκε πριν από 7-8 χρόνια, και ταυτόχρονα η δημόσια διοίκηση ε, προβαίνει στην καθυστερημένη απληρωμή απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε βέβαια αυξήνεται ακόμα περισσότερο αυτό το crunch. Ε, και, ε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ε, η σωστή διαχείριση είναι κάτι το οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που θέσατε. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη έχουμε έναν τραπεζικό τομέα στον οποίο υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες και σε ορισμένες χώρες ε, οδηγούμαστε ακριβώς σε αυτήν την εξάλληψη αν θέλετε της υπερπροσφοράς τραπεζικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν αυτή η ενοποίηση με την έννοια δηλαδή, των συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζών θα μπορούσε να έχει κάποια χρησιμότητα έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τραπεζών. Πάντως, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκείνο που θα θέλαμε να δούμε είναι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, διασυνορική ενοποίηση του τραπεζικού τομέα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε παρατηρήσει κατά τελευταία χρόνια είδαμε ορισμένες τέτοιου είδους ε, σχονεύσεις, δηλαδή κάποιες συμφωνίες μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας, αλλά ε, πέραν αυτών των ε, επιμέρους περιπτώσεων δεν είδαμε κάτι ως ευρύτερο φαινόμενο. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια τραπεζική ένωση, τότε πραγματικά τότε χρειαζόμαστε να υπάρχουν και πραγματικές ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή που υπάρχουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και θα επιτρέψει πράγματι την σωστή ύπαρξη μια ενιαία αγορά για τι τράπεζε. Τέλο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη διαφάνεια που θέσατε, συμφωνούμε πλήρω ότι δηλαδή πραγματικά η ανάληψη, το ευθυνό, το accountability και το καταξύ παίζουν ε, ζωτική σημασία. Αλλά ε, σε ό,τι αφορά το CSPD και στο συγκεκριμένο ζήτημα που εξετάζουμε, να σα πω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει στρέβλωση στην αγορά. Δηλαδή δημοσίευση. Οπότε θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες ε, ε, αρνητικές συνέπειες. Γνωρίζετε ποια είναι η δική μας στάση, ποια είναι η δική μας οπτική γωνία και ποια είναι η πολιτική μας. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε δημοσιεύσεις γιατί αυτής δηλαδή της, ε, αυτού του, του target, γιατί ακριβώς θα μπορούσαμε ακριβώς να υπονομεύσουμε τα αισθήματα διαφάνειας και, για του συγκεκριμένου κρατούς Πολύ ωραία. Δεν έχουμε διασυνοριακές ε, ε, συγχωνεύσεις γιατί υπάρχουν κίνητρα, ρυθμιστικά αντικίνητρα και γι' αυτό δεν προχωράει και η Τραπεζική Ένωση ε, και έχουμε μπλακεί και εγκλωβιστεί σε αυτό τον κύκλο που ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τον διαρρήξουμε έστω στην επόμενη θητεία. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση να θέσω μια ερώτηση που αφορά στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή κατά πόσον μπορεί και αυτή να συμβάλλει στη σταθερότητα των τιμών. Κάτι που είναι βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τους τελευταίους μήνες διαπιστώσαμε ότι μειώνεται το ποσοστό του πληθωρισμού, φτάνει περίπου στο 2% και γι' αυτό το λόγο έχουν επιβραδυνθεί και οι νομισματικές πολιτικές. Σήμερα όμως ε, διαπιστώνουμε ο πληθωρισμός του Μαρτίου φτάνει στο 1,4%. Σήμερα το πρωί το διαβάσαμε αυτό και πολλοί προβλέπουν ότι θα αποτύχει πλήρως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ με την έννοια ή στο βαθμό που δεν θα μπορέσει να επιτύχει το στόχο του πληθωρισμού που είναι να κυμαίνεται γύρω στο 2%. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την αναχρηματοδότηση ε, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εσείς δεν θεωρείτε ότι θα μπορούσε ε, να υπάρξει και μία περίοδος quantitative easing με την έννοια ότι όσον αφορά την ποσοτική χαλάρωση αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις προοπτικές για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ε, είδα λιγάκι το θέμα της εξέλιξης του πληθωρισμού και ε, τα κίνητρα του πληθωρισμού. Αν δούμε λιγάκι τον επίσημο πληθωρισμό, ε, θα διαπιστώσουμε ότι οι ενεργειακές τιμές ε, άσκησαν τεράστια επιρροή και αυτό είναι το βασικό αίτιο, γιατί υπήρξε αυτή η επιβράδυνση του πληθωρισμού, η μείωσή του στο 1,4% που δεν είναι ακριβώς ο στόχος μας, απέχει λιγάκι από το στόχο μας που είναι, σας είπα, πάνω κάτω γύρω στο 2%. Όσον αφορά τώρα τον υφέρποντα πληθωρισμό, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ο υφέρπον πληθωρισμός είναι ένα σταθερό στοιχείο του πληθωρισμού και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στον υπολογισμό του μέλλον, της εξέλιξης του πληθωρισμού στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιβράδυνση από ένα και κάτι πήγαμε στο 0,8%. Εγώ νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην ε, ύφεση της οικονομίας. Αν υπάρξει ανάκαμψη των οικονομικών δραστηριοτήτων προς το τέλος του έτους, αυτή είναι η πρόβλεψη που έχουμε εντάξει στις ετήσιες ε, προβλέψεις μας του 1,4%. Αλλά αυτό που προβλέπουμε είναι ότι το πρώτο εξάμεινο του έτους θα έχουμε οικονομική ύφεση και μετά η οικονομία θα ανακάμψει κατά το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Ε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να αυξήσουμε και πάλι τον υφέρποντα πληθωρισμό. Παράλληλα, όσον αφορά την, ε, νομισματική προσαρμογή, έχουμε προσφέρει ρευστότητα, άπλετη ρευστότητα, οι ε, χρηματοδοτικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις που και οι δύο ε, χαίρουν και απολαμβάνουν ε, πολύ καλές συνθήκες τόσο όσον αφορά τα επιτόκια όσο και τη διαθεσιμότητα κονδυλίων και δανείων. Άπλετη λοιπόν ρευστότητα, πολύ καλούς όρους δανειοδότησης. Αυτά υπάρχουν και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν. Παράλληλα βέβαια υπάρχει και το θέμα της εξέλιξης των μισθών. Γνωρίζετε ότι εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό το τι θα συμβεί. Γιατί βλέπουμε ότι αυξάνονται κατά 2 περίπου 0,5% σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες η εξέλιξη είναι ακόμα μεγαλύτερη, η αύξηση των μισθών. Ε, η αύξηση λοιπόν των μισθών διαρωτώμεθα γιατί αυτή δεν αντανακλάται στον υφέρποντα πληθωρισμό, στον επίσημο πληθωρισμό και στις ε, τιμές ελιανικής. Εκεί υπάρχουν πολλές ε, εξηγήσει. Ίσως να οφείλεται στην κρίση, ίσως να οφείλεται στις διαρθρωτικές αλλαγές των αγορών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Κατά το παρελθόν ε, ήταν διαφορετική η κατάσταση σε σύγκριση με τώρα. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα, νομίζω ότι έχουμε ε, πολλά εναλλακτικά εργαλεία. Στο τελευταίο Συμβούλιο αποφασίσαμε ε, να εισάγουμε ένα καινούριο στοιχείο TLTRO, το υπαριθμόν 3, Πρόκειται για τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροχρό... μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Αυτά θα κρυθούν κατά τις επόμενες εβδομάδες ε, και θα συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα θετικοί όσον αφορά τη χρηματοδότηση τραπεζών έτσι ώστε να ελέγχεται το τραπεζικό κόστος ε, και να υπάρχει μια ήπια νομισματική πολιτική. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι αναβάλουμε λιγάκι την ημερομηνία όπου θα αυξηθούν λιγάκι τα επιτόκια και αυτό το μεταθέτουμε προς τα τέλη του έτους ή ακόμα και αργότερα. Μπας περιπτώσει, όλες οι αναλλακτικέ λύσεις είναι ανοιχτές. Αν συμβεί κάτι το περίεργο, αν δούμε το χάρη ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος μας, ε, ε, δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας και για να το πετύχουμε ε, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στο οπλοστάσιό μας. Ευχαριστώ. Στέφαν. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Ευχαριστούμε για την εισαγωγική σας παρουσίαση. Είχα μια πρώτη ερώτηση που με καλύψατε όμως για τα επιτόκια. Και έχω λοιπόν δύο σύντομες ερωτήσεις μόνο. Η πρώτη, ε, τις ανισορροπίες στόχου 2. Μετά από μια φάση όπου η, το κενό ισορροπίας των στόχων 2 ε, μειώθηκε, τώρα αυξήθηκε. Αυτό απασχολεί την έκτα. Και αν ναι, Έχετε κάποιο εργαλείο για να αντισταθμίσετε αυτή την τάση και το δεύτερο ερώτημα αφορά τον Brexit. Υπάρχει κάποια συζήτηση με την Τράπεζα Αγγλίας για να μετριαστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του Brexit. Uh, on target. Για την πρώτη ερώτηση. Η αύξηση του χάσματος για το στόχο 2 έχει να κάνει με την αποκεντρωμένη εφαρμογή του προγράμματος APPP, αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Αυξήθηκαν έτσι τα χάσματα ανάμεσα στις ε, διάφορες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση στους πιθανούς φόβους για το τι θα συμβεί όπως συνέβη ας πούμε, στη μέση της κρίσης. Τώρα έχει να κάνει περισσότερο με κάποια λειτουργικά θέματα λόγω της συγχρονισμένης ή μη συγχρονισμένης εφαρμογής του προγράμματος APP. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας τη φάση της καθαρής αγοράς περιουσιακών στοιχείων, θα δείτε στο εγγύς μέλλον ότι αυτές οι αποκλήσεις, αυτά τα χάσματα θα μειώνονται και θα έχουμε ε, μία σύγκληση σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς των διαφόρων ε, χωρών. Για το Brexit. Είπα ότι οι συνέπειες ενός no deal, απουσία συμφωνίας, είναι διαχειρίσιμες. Αλλά δεν θα είναι αμελητές. Γιατί είναι διαχειρι... Ε, διαχειρίσιμες γιατί τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι διοικητές των τραπεζών έχουν λάβει αποφάσεις για να μειώσουν τις πιθανές συνέπειες ενός no deal που είναι το χειρότερο σενάριο, όπως ξέρετε πολύ καλά. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο προετοιμασμένος για ένα Brexit χωρίς ε, συμφωνία, για ένα no deal Brexit, σε σχέση με το πώς ήταν πριν έξι μήνες. Το πρόβλημα ε, δεν είναι μόνο ότι είναι όμως διαχειρίσιμο, αλλά δεν θα είναι αμεληταίο απ' την άλλη. Γιατί? Γιατί οι αγορές δεν έχουν τιμολογήσει την πιθανότητα ενός σενάριου no deal. Δεν έχουν αποτιμήσει αυτή την πιθανότητα. αν συμβεί το no deal, ας πούμε, το χειρότερο σενάριο. Γιατί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, έτσι. Για να... Και θα αντιμετωπίσουμε πιο άνετα κάτι πιο εύκολο. Ε, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, καταρχάς υπάρχει μια επιβράδυση της οικονομίας. Και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διαμορφώνουν έτσι την οικονομία που τους ανέφερα πριν. Ένα no deal το οποίο δεν έχει αποτιμηθεί 100% από τις αγορές και στο οποίο ας πούμε αποδίδουν χαμηλή πιθανότητα να συμβεί. Η, δηλαδή no deal ή μη συντεταγμένη αποχώρηση ας πούμε του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μπορούσε λοιπόν αν συμβεί κάτι τέτοιο να μεγιστοποιήσει τις αρνητικές τάσεις που υπάρχουν λόγω της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μπορεί να επηρεάσει λοιπόν. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για τα, την επίπτωση ε, των CCP, των παραγόγων. Μπορεί να επηρεάσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα, το συνέστημα και αυτό μπορεί να ε, μεγιστοποιήσει τα αρνητικά στοιχεία που βρίσκονται, που υποκρύπτονται πίσω από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επομένως, ένα Brexit με no deal, χωρίς ε, συμφωνία, σίγουρα δεν είναι κάτι αμιλητέο. Πρόεδρος. Ο κύριος Φερνάνδης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι που είστε εδώ και εξετάζουμε μαζί τη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την, το feedback, τη δουλειά που έκανε μετά τις, τις συστάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας ήταν διαχειριστές της επικοινωνίας. Πολύ επιδέξει διαχειριστές. Ε, ε, ε επικοινωνούσαν για την νομισματική πολιτική. Με στόχο την ε, υλοποίηση των στόχων της τράπεζας και την επίτευξη του στόχου του 2%. Τις τελευταίες όμως εβδομάδες παρατήρησα ότι υπάρχει κάποια σύγχυση στον τρόπο που επικοινωνεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καταρχάς, εντόπισα ότι μετά την τελευταία συνεδρίαση στο βαθμό που η νομισματική πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί και οι προοπτικές ε, ανάπτυξης και πληθωρισμού μετριάζονται, είναι λογική η ανακοίνωση της τράπεζας για να αυξηθεί η ρευστοποίηση τους ε, επόμενους μήνες. Και βλέπουμε ε, μία επιβράδυση της δραστηριότητα και του πληθωρισμού. Μετά λοιπόν από την επίσημη ανακοίνωση της ε, Κεντρικής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΕΚΤ ανακοίνωσε την πιθανότητα αναθεώρησης των αρνητικών ε, επιτοκίων στις καταθέσεις ε, των τραπεζών και στον ισολογισμό της ΕΚΤ. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι σε ποιο βαθμό τη μία εβδομάδα χρειαζόμαστε περισσότερη ρευστότητα για να διατηρήσουμε ας πούμε την νομισματική πολιτική την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα θέλετε να αναθεωρήσετε τα αρνητικά επιτόκια, ούτω ώστε να λάβετε ε, αντίθετη απόφαση σε σχέση με αυτή που είχατε λάβει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η αναθεώρηση των διαφόρων αρνητικών επιτοκίων είχε αποφασιστεί ήδη από την ΕΚΤ και σε ποιο βαθμό αυτή η αναγγελία θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στην επικοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται την νομισματική πολιτική ως κεντρική τράπεζα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας ε, διευκρινίσω κάτι. Όσον αφορά την ανακοίνωσή μας ε, και την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες, επ' αυτού τι έγινε. Αποφασίσαμε να μην δεχτούμε καμία αλλαγή στα επιτόκια. Αποφασίσαμε να αναβάλουμε μέχρι το τέλος του έτους. Αποφασίσαμε λοιπόν αποφασίσαμε να αναβάλουμε τις εξελίξεις ε, και γι' αυτό το λόγο εφαρμόζουμε μια πιο προσαρμοσμένη νομισματική πολιτική όπου βεβαίως ε, αυτό συνοδεύτηκε και με την εισαγωγή του TLTRO 3 δεχτήκαμε να αναβληθούν κάποιες άλλες διαδικασίες τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 2021. Όλη η ανακοίνωση λοιπόν δική μας ήταν κάτω από αυτό το πρίσμα. Ήταν με αυτή την έννοια. Ήταν η αντίδρασή μας στην επιβράδυνση της οικονομίας, στην επιβράδυνση του πληθωρισμού. Ως εκ τούτου τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2019 δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των αρνητικών επιτοκίων. Απολύτως καμία αύξηση. Εδώ το θέμα που τίθεται είναι το εξής. Κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να αποφύγουμε, να επιβάλλουμε αρνητικά επιτόκια στις ε, τράπεζες και στις καταθέσεις που έχουν οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι κάτι που και αυτό δεν έχει συζητηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ούτε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως άλλο θέμα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι θα συνεχίσουμε να αναλύουμε τις ε, δυνατότητες ε, που υπάρχουν γιατί υπάρχουν και διαφορετικές ε, νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται. Μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση, γιατί δεν είχαμε και αυτή τη συζήτηση ε, ούτε στο εκτελεστικό γραφείο της ΕΚΤΟ, ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα βασικά όργανα της ΕΚΤΟ. Ο κύριος Γκέρολτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση ε, συμπληρωματική που αφορά στο Brexit. Ε, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν ιδιαίτερα ειλικρινής και ουσιαστικός της απαντήσεις Όσον αφορά το θέμα της ισοτιμίας ανάμεσα στη Βρετανική Λίρα και το Ευρώ. Μέχρι τώρα και κυρίως μετά την πρώτη ψηφοφορία για το Brexit στο Κοινοβούλιο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, θα περίμενε κανείς ε, υποτίμηση της Βρετανικής λίρας σε σχέση με το ευρώ. Πράγμα που δεν συνέβη προς έκπληξή μας, γιατί περιμέναμε ακριβώς το αντίθετο. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι τελικά, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τελική αποτίμηση και ρωτώ, εσείς θεωρείτε ότι θα αποδυναμωθεί η λίρα σε σχέση με το ευρώ μετά την ε, ε, τελική συμφωνία που ενδεχομένως να είναι αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Ίσως εσείς ε, να είστε καλύτερα ενημερωμένοι από μένα. Εγώ λυπάμαι, ε, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι είδου αποχώρηση της μεγάλη Βρετανίας ε, θα έχουμε εν το χρόνο. Δεν θα τολμούσα ποτέ να πω τι θα συμβεί, δεν ξέρω τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Μπα περιπτώσει, αυτό, αυτή η λύση, αυτό το σενάριο ε, της μη συμφωνίας, αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συζητιέται στις αγορές, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα συμβεί, είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να προκύψει, οι αγορές προφανώς θα αντιδράσουν. Οι αγορές αντιδρούν, αυτό είναι μια πραγματικότητα κυρίως ε, αν τελικά αυτό που θα προκύψει δεν θα είναι το αναμενόμενο σενάριο. Οι αντιδράσει θα μπορούσαν να ποικίλουν. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, ε, να υπάρξουν επιρροέ στην ισοτιμία, στα σπρέντε, σε οτιδήποτε. Για μένα αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι ακριβώς το θέμα το πώς θα εξελιχθεί η ισοτιμία λίρας ευρώ. Το κέριο ερώτημα είναι ότι βεβαίως και θα υπάρξουν ε, πολύ αρνητικές ε, εξελίξεις. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή η αποχώρηση χωρίς συμφωνία επειδή έχουμε και κάποια ε, ευαίσθητη οικονομία αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια εφεσιακή τάση, ίσως αυτός ε, θα μπορούσε να είναι άλλος ένας παράγων, ο οποίος θα δυσχεράνει την ανάκαμψη της ε, οικονομικής δραστηριότητας που εμείς προβλέπουμε ότι θα προκύψει κατά το δεύτερο εξάμεινο του έτους. αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ακριβέστερες προβλέψεις. Οι αγορές ε, δεν ε, ε, έχουν αυτή τη στιγμή αντιδράσει και δεν έχουν πει τίποτα σχετικά με την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Η κυρία Περές. Στην ετήσια έκθεσή σα, την οποία μόλι ανακαλύψαμε, μιλάτε για τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εφαρμόσει διάφορα κριτήρια. Στην κοινή γνώμη υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για το πώς η νομισματική πολιτική λαμβάνει υπόψη τους στόχους του μείον δύο ε, βαθμοί Κελσίου, δηλαδή, τη Συμφωνίας του Παρισιού. Στο πρόγραμμα αγορά σα ή εξαγοράτη η εφαρμογή μία στρατηγικής για το μείον δύο βαθμοί Κελσίου, δεν έχει προωθηθεί σημαντικά και στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, τουλάχιστον υπάρχει μια ολόκληρη πολεμική για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε μια στρατηγική αντίθετη με τους στόχους ε, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση, θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχετε κάνει τη χρονιά που μας πέρασε σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για το προσωπικό. Υπάρχει ένα ανισχυτικό ερώτημα για τις συνθήκες διαπραγμάτευσης των κοινωνικών όρων και των κοινωνικών συνθήκων και ε, το θέμα της βελτίωσης της διαχείρισης, της διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας να ξεκινήσω με την κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή θα πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικά ταμεία, σε όλους, ότι η κλιματική αλλαγή εάν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, θα αποτελέσει έναν σημαντικό διαρθρωτικό κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα πρέπει δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε τις τράπεζες προκειμένου να αντιληφθούν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράγοντα που θα δημιουργήσει ακριβώς νέες προκλήσεις και νέους κινδύνους αποσταθεροποίησης. Καταρχήν, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ναι, αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα η κλιματική αλλαγή. Αλλά ε, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στις τράπεζες ε, και γενικότερα σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Νομίζω πως ε, υπό κανονικέ συνθήκε, όταν εφαρμόζουμε την δική μα εκτίμηση σε ό,τι αφορά του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, μέχρι στιγμή δεν λαμβάνουμε υπόψη μα την κλιματική αλλαγή. Αλλά τώρα θα αρχίσουμε να την συμπεριλαμβάνουμε σε αυτέ τι εκθέσει μα. Όπω θα αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε, για παράδειγμα, και το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων, που δηλαδή θα αποτελέσει και αυτό παράγοντα δυνητικό απεσταθεροποίηση, όπω θα αναφέρεται στι εκθέσει μα. Άρα λοιπόν θα αρχίσουμε ακριβώς να ε, βλέπουμε, να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή ως ε, παράγοντα δυνητικής, ακριβώς διαρθρωτικής χρηματοπιστωτικής αποσταθεροποίησης. Αυτό λοιπόν θα γίνεται λόγω και πιο ορατό από τη δική μας πλευρά ως ε, εποπτική αρχή, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ε, αρχή αρμόδια για την παρακολούθηση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Άρα λοιπόν αυτή η πτυχή θα περιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο στι δικέ μα ε, αξιολογήσει και στι δικέ μα εκθέσει θα εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο στο πλαίσιο ε, των δυνητικών ακριβώ απειλών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη της μεταξύ των δύο φύλων, τη ισότητα των δύο φύλων, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά δυστυχώ έχουμε αυτή την κατάσταση που ισχύει σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και ελπίζουμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξουν κάποιες ε, αλλαγές εκεί της φρουράς αν θέλετε, έτσι ώστε ακριβώς να έχουμε πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φίλων στο ε, Συμβούλιο. Το εκτελεστικό, αν θέλετε, συμβούλιο, το ε, Executive Board. Αλλά και γενικότερα στο προσωπικό, στο σύνολο του προσωπικού της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να να διασφαλίσουμε ακριβώ αυτή την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Ε, γιατί θεωρούμε πω είναι σημαντικό ε, παράγοντα ε, για την ποικιλομορφία μα. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Τρεμόζας, ο κύριο Μάου στο πλαίσιο τη Διαδικασία Κατσδιά. Για ένα λεπτό. Ναι, σε ό,τι αφορά τι απαντήσει που μου έδωσε ο κύριο Εντεκίνητο σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη διαφάνεια. σω εγώ λοιπόν να μην εξέφρασα σωστά αυτό που ήθελα να πω γιατί ο κύριο Ντεκίντος μου είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφεύγει να δημοσιοποιεί ε, τις ε, επωνυμίε των επιχειρήσεων προκειμένου να αποφύγει επιπτώσεις στις αγορέ. Όμως ε, πριν από δύο χρόνια, λόγω ακριβώς των πιέσεων που ασκήθηκαν από τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβησε ακριβώς την δημοσιοποίηση των holding CSPP. Ε, Οπότε θεωρώ πως θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια καλή απαρχή, ένα καλό παράδειγμα. Ε, και σίγουρα αυτό επειδή θα προκύψει και στην επόμενη βουλευτική περίοδο, καλό θα ήταν να το θίξουμε. Κύριος Δεκίδε. Ναι, ε, έχετε δίκιο. Δημοσιοποιήσαμε τις απονομίες αυτών των επιχειρήσεων, αλλά δεν δημοσιοποιήσαμε πολλές άλλες πληροφορίες. Ε, δηλαδή για παράδειγμα ο βαθμός εξέτασης ε, την οποία, στον οποίο υποβάλαμε την κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας ε, Ντεγκίντος για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Δυστυχώς στο πλαίσιο αυτής της προεκλεγικής περίοδου λοιπόν έχουμε αυτή την χαμηλή προσώπηση από του συναδέλφου. αλλά παρόλα αυτά η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σα ευχαριστούμε και εσά προσωπικά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Θα διακόψουμε πολύ σύντομα τις εργασίε μα. γιατί πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών πρωτού περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερής σα διαταξής. Οπότε θα διακόψουμε για 10 λεπτά.